ε, όπου έλαβα μια αντίρρηση από την ομάδα EFTD προς τη σύσταση της επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, ώστε να μην φέρουμε αντίρρηση στην, ε, ε, στον κανονισμό της Κομισιόν 2 Οκτωβρίου 2014 όσον αφορά το προσωρινό σύστημα δόσεων στις συνεισφορέ που θα καλύψουν τα διοικητικές δαπάνε του Συμβουλίου το νέο Συμβουλίου Εξυγίαση, σύμφωνα μάλλον κατά τη διάρκεια τη προσωρινής Διαδικασία. Κατά συνέπεια θα ψηφιστεί η σχετική σύσταση. Η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών θα είναι η Τετάρτη 10 το πρωί και η προθεσμία για χωριστέ ε, ε, ψηφοφορίε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ και τώρα συνεχίζουμε τη συζήτηση για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών και δίνω το λόγο στην κυρία Χιμένα Μπεσερέλ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Από τότε που ήρθα εδώ στο Κοινοβούλιο, η περάσπιση των θυμάτων ε, ήταν προτεραιότητά μου και όπου και αν είμαι θα είναι προτεραιότητά μου. Οι γυναίκες στην Ευρώπη, τα θύματα βίας μας ζητούν να μιλήσουμε με μία σαφή φωνή και να ενώσουμε